Uh, good afternoon, colleagues. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιστεύω να έχετε ξεκουραστεί και να έχουμε μια καλή παραγωγική νέα σεζόν. Κάθε επιτυχία για όλους και όλες μας λοιπόν σε αυτή την περίοδο που μόλις ξεκίνησε. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 1 της Μέσιας Διάταξης, έγκριση του σχεδίου Μέσιας Διάταξης. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, προτείνω να εγκριθεί το σχέδιο Μέσιας Διάταξης. Δεύτερο σημείο είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 20 Ιουνίου. Σχόλια δεν υπάρχουν. Εγκρίνονται λοιπόν. Επόμενο σημείο. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Σε ό,τι αφορά τι συστάσει των συντονιστών τη 12η Ιουλίου. Αποφάσισαν λοιπόν στη συνάντησή του οι συντονιστέ ότι το θέμα τη Διεθνού ημέρα για τι γυναίκε του 2018 θα είναι συμμετοχή και πρόσβαση των γυναικών ε, στα μέσα ενημέρωση και τεχνολογίε πληροφοριών και επικοινωνιών και πώ επηρεάζουν και πώς μπορούν να αποτελέσουν μέσο για την ανέλυξη και τη χειραφέτηση των γυναικών. Επίσης, ό,τι αφορά την υλοποίηση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Άλτε θα αναλάβει την θέση για τις τροπολογίες και σε ό,τι αφορά τη σύσταση προς Συμβούλιο για τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για την 62η Σύνοδο της ε, Συνόδου του ΟΗΕ, η Γκουε και η Άλντε η κυρία Κοσλόφσκα και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ επίση παίρνουν εντολή να συμμετάσχουν στην ακρόαση που οργανώνει το UNDP στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2017. Το επόμενο σημείο τώρα τη μερσιά διάταξη είναι το σημείο 4, εργαστήριο με θέμα την αύξηση τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Έχει διοργανωθεί από το θεματικό τμήμα ΓΑΜΑ. Στην σημερινή μα συνεδρία, στο σημερινό εργαστήριο, θα καλωσορίσουμε καταρχάς ε, την εκπρόσωπο του πολιτικού γραφείου της ε, κυρίας Γιούροβα, την κυρία Μόνικα Λατουμάνοβα, που θα μας μιλήσει για τις προτάσεις της Κομισιόν και συγκεκριμένα την οδηγία για την εξορόπηση, για την συμφιλίωση οικογενειακού και οικογενειακού, οικογενειακού επαγγελματικού βίου. Και έχουμε και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, ε, την καθηγήτρια Μπούρη, τον δόκτορα Τίμο Άντιλα, θα μας μιλήσουν για τις προκλήσεις και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά και τα διαφορετικά ωράρια και τις προκλήσεις για την ε, συμφιλίωση της ε, επαγγελματική και οικογενικής ζωής και η κυρία Δαβάκη θα μας μιλήσει για τα απορίσματα της μελέτης για την ε, δημογραφία και τις οικογενικές οικογενειακές πολιτικές. Κυρία Μόνικα Λαντμάνοβα καταρχάς θα πάρει το λόγο από το πολιτικογραφείο της Επιτρόπου Βέρα Γιούροβα. Έχετε 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Όπως είπε και η Πρόεδρος, έχω έρθει εδώ για να επανεπιβεβαιώσω τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε όλοι και όλες την κατάσταση και τη σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει ισότητα. Ξέρουμε ότι ε, υπάρχει ε, εκπροσώπηση των γυναικών ακόμη στην αγορά 65% ε, για τις γυναίκες και 75% για τους άνδρες τα επίπεδα, τα ποσοστά απασχόλησης. Χάνονται ταλέντα, χάνονται πόρια την κοινωνία γιατί αποφυτούν από πανεπιστήμια γύρω στο 6% γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Και όπως τα έλεγε η κυρία Γιούροβα, έχουμε τις πιο καλά, τις πιο μορφωμένες νοικοκυρές στην Ευρώπη. Όμως αυτό συνιστά στοχεία της αγοράς. Και δεν έχει νόημα δεδομένων και των κοινωνικών ε, καταστάσεων, ε, συνθήκων, μειώνεται, συρρυκνούται και δημογραφικά η κοινωνία. Από το 2008 το ποσοστό απασχόληση των γυναικών αυξήθηκε πολύ λίγο και υπάρχουν και οικονομικές απώλειες γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Τεράστια προβλήματα δημιουργούν αυτά, τα νούμερα τα ξέρετε 370 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Ευρώπη, 2,8% του ΑΕΠΑ. Και αυτό βέβαια αποτελεί απώλεια και για το δημόσιο προπολογισμό, δημόσια κονδύλια. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συνεχίζεται. Γνωρίζουμε επίσης ότι ζούμε σε καινούριου ε, καιρούς πολύ έκτακτους και διαφορετικούς ό,τι αφορά τα ε, ωράρια και τον τρόπο εργασίας. Έχουμε νέα μοτίβα, νέα τρόπους εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν ε, τα καθήκοντα των εργαζομένων να μπορούν να συμφιλώνονται με τα καθήκοντα κατοίκων. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αλλαγών αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταθέσει μια νέα σύγχρονη πολιτική για τη συμφιλίωση της ε, οικογενειακή και επαγγελματική ζωής, για του εργαζόμενου γονεί και για όσου ε, φροντίζουν κάποιο μέλο τη οικογένειας. Στόχος μας μεταξύ άλλων είναι να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στις οικογένειε, κάτι πολύ σημαντικό δεδομένου των δημογραφικών εξελίξεων. Αυτή είναι η άποψή μου. Η νέα πολιτική λοιπόν θα πρέπει να ενθαρρύνει να υπάρχουν σύγχρονες διευθετήσεις, να είναι σύγχρονες οι δομές έρημνας και να μπορεί έτσι η οικογένεια να μπει στην αγορά εργασίας και να δοθούν τα απαιτούμενα κίνητρα. Το Eurofound προβλέπει τη συμμετοχή των γυναικών και το πώς θα αλλάξει αυτή με βάση το αν θα γίνουν παρεμβάσεις ή δεν θα γίνουν παρεμβάσεις. Και το αποτέλεσμα της μελέτης είναι ότι με συστηματική συντονισμένη δράση που θα στηρίζει τις γυναίκες στην αγορά εργασίας θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και στην οικονομική κατάσταση των γυναικών αλλά και στο κοινωνικό πλαίσιο. Διότι τα άτομα που είναι στην αγορά εργασίας τείνουν να θεωρούν ότι έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής. Αξιολογούν την ποιότητα ζωής τους ε, με πιο θετικό μάτι σε σχέση με όσους είναι εκτός αγοράς εργασίας. Άρα, δείχνει η μελέτη αυτή πως πρέπει να ακολουθήσουμε μια σωστή πολιτική για να ελκύσουμε τις γυναίκες ε, στην αγορά εργασίας και θα πρέπει ταυτόχρονα να δώσουμε κίνητρα και στους εργοδότες. Να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση για εργατικό δυναμικό και σε ό,τι αφορά τις, ε, τα ευέλικτα ωράρια και την ε, οργάνωση του χρόνου εργασίας πρέπει να είναι πιο ελαστική. Δέκα μη νομοθετικές δράσεις και μια νομοθετική δράση προ την Κομισιόν, που αλληλοενισχύονται. Και με το συνδυασμό των δύο θα φέρουμε αυτή την επιδιωκόμενη αλλαγή, όπως προείπα. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνουμε νέες σύγχρονες ε, διευθετήσεις για τις άδειες. Να έχουμε επίσης καλύτερη πρόσβαση και βελτίωση των ε, υπηρεσιών μέρημνας, φροντίδας, και να μπορεί ο δεύτερος γονιός ε, να βρει και αυτός δουλειά. Να καταργηθούν τα αντικίνητρα και στηρίζουμε τα κράτη-μέλη στις προσπάθειες που καταβάλουν στο ζήτημα της οικογενειακής πολιτικής, λαμβάνοντας το κοινωνικό υπόψη, το κοινωνικό και δημογραφικό πλαίσιο. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του την ε, ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Και στόχος πολιτικής είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. για να λαμβάνονται υπόψη ε, και ε, οι κοινέ ευθύνε και τα, οι παροχές να είναι σχεδιασμένες με βάση την ισότητα των φίλων. ο πατέρας περνάει περισσότερο καιρό με το παιδί του, θα έχει και καλό, καλύτερη σχέση μακροπρόθεσμα με το παιδί. Αλλά και θα φανεί ότι δεν χάνει τις γονικές του αρμοδιότητες, αλλά αναλαμβάνει και τις ευθύνες του νοικοκυριού. Θα είναι ένας πραγματικός τηλοβάτης της οικογένειας. Και από δημοκρατική πλευρά θα είναι θετικό αυτό. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε αποφασίσει είναι να τροποποιήσουμε την οδηγία για τη γονική άδεια, διατηρώντας τη φυστάμενα δικαιώματα, αλλά βελτιώνοντα αυτά τα δικαιώματα και προσθέτοντα άλλα. Βελτιώνοντα τα δικαιώματα των και των γυναικών, εισάγουμε και νέε παροχέ. Η μία για αφορά του ε, γονεί νεογέννητων, να παίρνουν δηλαδή πατρική άδεια, ε, άδεια πατρότητα, και για ρυθμίσεις για όσους έχουν προστατευόμενο εξαρτώμενο μέλος. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι μη νομοθετικές δράσεις όπως είπαμε, 10 τον αριθμό για την άδεια, για να μην υπάρχουν διακρίσεις, για να μην υπάρχουν απολύσεις, για να αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια των δομών φροντίδας και τα φορολογικά αντικίνητα. Ταξί αυτών των νομοθετικών δράσεων περιλαμβάνει τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Να τις ενθαρρύνουμε θέλουμε ώστε πολιτικές ευεξίας να εισαχθούν για τους εργαζομένους ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη ένα ελαστικό ωράριο ή ε, δομές φροντίδας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ άλλων μια πλατφόρμα για την ε, παρουσία των καλών πρακτικών. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα για τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για να παρακολουθούμε ποιε είναι οι ανάγκε και να μπορούμε να αντιδρούμε με βάση την παρακολούθηση αυτή, επαναπρογραμματίζοντα την ε, υφιστάμενη χρηματοδότηση και επενδύοντα στι υποδομέ. Θέλουμε επίση να εστιάσουμε εκ νέου ε, τη χρηματοδότηση και του Ταμείου Juncker ώστε να στηρίζουν τα κονδύλια αυτά τις κοινωνικές επενδύσεις περισσότερο. Τέλος, θέλουμε να εστιάσουμε και στις φορολογικές πολιτικές. Να δώσουμε καθοδήγηση για την προσαρμογή των πολιτικών αυτών, ώστε να μην είναι ευεργετικέ μόνο για έναν, ε, τον ένα γονέα, ο οποίος φέρνει το εισόδημα στην οικογένεια, αλλά να ενισχύσουν και τον δεύτερο γονέα. Με αυτή την σέγγιση, με αυτή τη σύγχρονη πολιτική, χαράσουμε το δρόμο για τον 21ο αιώνα. Δεν θα γίνει μια ανοιχτή αλλαγή, το γνωρίζουμε. Όπως γνωρίζουμε ότι χρειάζονται δύο ε, για να, να το ταγκό, όπως λένε στα, στα αγγλικά. Βλέπουμε επίσης ε, η νέα γενιά, ιδίως οι άντρες, ε, να ενδιαφέρονται περισσότερο ε, και πρόσφατα ε, είχαμε μια συνέντευξη του πρόεδρου της λιθανικής ε, ομάδας μπάσκετ. Την ευχαριστήθηκα πολύ αυτή τη συνέντευξη που μίλησε εκεί για τα παιδιά και για την άδεια πατρότητα, Είναι ο γνωστός μπασκετπολίστας για Kaip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 The Ήταν ένα βίντεο YouTube. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το δείτε και από μόνοι σας. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ Η Επιτροπή μας ε, δουλεύει συστηματικά και συνεργάζεται με την Επίτροπο Γιούροβα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το πακέτο για τις νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις και ελπίζουμε να τις επεξεργαστούμε περαιτέρω. Με εξέπληξε η απόφασή σας να επιλέξετε αυτόν τον Λιθουανό διάσημο μπασκετμπολίστα, ο οποίος είναι σε μια λιθουανική ομάδα μπάσκετ. Και μας έδωσε μια πολύ λογική, πολύ ανθρώπινη εξήγηση για το πώς ένας πατέρας πρέπει επίσης να συμμετέχει στην ε, ανατροφή των παιδιών του. Ήταν πολύ ε, βιωματική αυτή η αφήγηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ελπίζω πολύ να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα. Ο παίκτη αυτός λοιπόν είναι ε, μοντέλο για τους συμπατριώτες μας. Και τώρα ο, η καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πρόσκληση και την πολύ συναρπαστική εισήγηση. Έχω κάποιες διαφάνειες, οπότε θα διακόπτω για να τις αλλάζω. Είμαι ανεξάρτητη εμπειρογνώμων, δεν εκπροσωπώ κανέναν. Είμαι συντονίστρια και στο σχετικό δίκτυο για την ισότητα των φύλων και τη μη διακριτική μεταχείριση στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό που ήθελα να κάνω σήμερα Ελπίζω ότι θα μπορώ μόνιμο με το remote να αλλάζω τις διαφάνειες, αλλά δεν μπορώ. Ε, η ισορροπία των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ισορροπία εργασίας προσωπικού βίου. Θα ήθελα λοιπόν να αποτιμήσουμε και την ισχύουσα νομοθεσία ε, για να δούμε τι ε, νόημα έχει η πρόταση και μετά θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην πράξη ε, και συγκεκριμένα στις κάτω χώρες, τι συμβαίνει στην Ολλανδία και πώς σκοπεύουμε να ενσωματώσουμε την οδηγία στην οδηγία μας. Επόμενο συμπεράσματα, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Όπως υπόθεκε προηγουμένως, Η ισορροπία επαγγελματικού και γονεϊκού βίου δεν αφορά μόνο τις άδειε. Έχει να κάνει και με τις, με τις υποδομές για την φροντίδα των παιδιών, με, τις, με τα φορολογικά κινήτρα και το καθεξής. Γι' αυτό χαίρομαι που είναι ευρύ το πακέτο. Και θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ στο πρώτο σκέλο, το κεκτημένο, το κοινωτικό κεκτημένο για την ισορροπία επαγγελματικού οικογενειακού βίου. Πολλά έχουν γίνει ήδη. Έχουμε την οδηγία αναδιατύπωση για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην απασχόληση αυτό περιλαμβάνει και την ε, ε, ακρεφνή διάκριση λόγω φύλου, η οποία έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλές πολλές υποθέσεις. Για παράδειγμα, η μη ανανέωση μιας σταθερής σύμβασης, εφόσον δεν είναι τεκμεριωμένη ε, και γίνει για λόγους εγκυμοσύνης, είναι άμεση διακρίση λόγω του φύλου και απαγορεύεται. Το αποφάσισε το δικαστήριο σε μια υπόθεση. Επίσης, η αποτροπή από την άμεση διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, λόγω, χάρη, λόγω της γονικής άδειας ή της εγκυμοσύνης. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση στο δικαστήριο ήταν ε, η Μπίλκα, η υπόθεση Μπίλκα. Επόμενη διαφάνεια, επί προσθέτως, έχουμε διατάξεις για την ε, επιστροφή από την άδεια έχει δικαίωμα να γυρίσει κάποιος ή κάποια στη δική του θέση και να έχει και βελτιώσεις εκεί. Επίσης για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. σε επίπεδο άδεια ασθενεία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 14 εβδομάδε αμοιβόμενε και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η απαγόρευση κατά τη αποπομπή ή απόλυση. Επόμενη, επόμενη. Από την αρχή της εγκυμοσύνης μέχρι το τέλος της ε, εγκυμοσύνης και της άδεια μετρότητας. Αυτό έχει ερμηνευθεί με πολύ αυστηρό τρόπο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επιπλέον υπάρχει οδηγία για την ε, γονική άδεια, η οποία δίνει δικαίωμα σε γονική άδεια τουλάχιστον τέσσερις μήνες, εκ των οποίων ο ένας δεν μπορεί να μεταφερθεί, ε, πρέπει να ε, εκχωρηθεί μέχρι το παιδί να φτάσει στα 8 έτη. Αφορά γέννηση, οθεσία και εκεί μιλάμε για ε, άδεια χωρίς αμοιβή. Εκεί θα αλλάξει τα πράγματα η οδηγία. Επίσης έχουμε τους αυτοπασχολούμενους, την οδηγία για τους αυτοπασχολούμενους, η άδεια μητρότητα σε αυτή την οδηγία είναι σημαντική υπό την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ε, ωφελήματα από την άδεια μητρότητα, τουλάχιστον 13 εβδομάδες, και να υπάρχει και πρόσβαση σε προσωρινή αντικατάσταση. Τέλος, ήθελα να αναφέρω την οδηγία ε, εργασίας μερικού χρόνου με σχετικά δύναμα δικαιώματα προ όφελο των ευνοϊκών, ελαστικών εργασιακών συνθήκων. Αυτό είναι το κεκτημένο. Τώρα, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οδηγία για την Ισορροπία Οικογενειακού και Επαγγελματικού Βίου θα προσθέσει όλα αυτά. Είναι το ερώτημα. Επόμενο, μερικές, μερικά σημεία για να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν σοβαρά κινήτρα για τους άντρε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τις άδειες. Οι άδειε δεν σχετίζονται μόνο με τη φροντίδα των παιδιών, αλλά και με τους ασθενείς ή εξαρτώμενους συγγενείς. Δύο νέες άδειες έχουν προβλεφθεί. Πρώτα απ' όλα η άδεια πατρότητας για τους πατέρες, επευκαιρία της γέννησης του παιδιού, άσχετα από το ε, έγγαμο ή συζυγικό καθεστώς, 10 ημέρες και μετά η συζυγικο καθεστως δεκα ημερες και μετα η αδεια για τους φροντιστές για όσους παρέχουν προσωπική περίθαλψη υποστήριξη σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σε περίπτωση εξάρτησης συγγενούς. Η άδεια των φροντιστών είναι πέντε ημέρες το χρόνο. Δύο νέες άδειες στην πρόταση αυτή. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με τη γονική άδεια. Πρώτον, θα είναι ένα ατομικό ονομαστικό μη ε, μεταφερόμενο δικαίωμα για τουλάχιστον τέσσερι μήνε. Οι τέσσερις μήνε δεν θα αλλάξουν ω προ το δυνατότητα να μεταφερθεί αλλά θα αλλάξει ε, και η ηλικία του παιδιού μέχρι τα 12 έτη και όχι πλέον 8. Θα μπορεί να είναι 12 το παιδί, με να ληφθεί άδεια μέχρι τα 12 και θα εκκρατάται από το κράτο μέλο αυτό. Επίση θα ανακληθεί οδηγία 2018. Ε, Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο θα υπάρχει πληρωμή του ε, ανάλογου εισοδήματο ε, στο ύψος της άδειας ασθενείας, στην περίπτωση της άδειας πατρότητας, της γονικής άδειας ή της φροντιστικής άδειας. Δεν υπάρχει αλλαγή εδώ, γιατί όλα αυτά ούτως ή άλλως είναι αμοιβόμενα. Επιπλέον, θα υπάρχουν ισχυρότερα ε, δικαιώματα συγγνώμη, για τα ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις. Μέχρι τα 12 έτη του παιδιού και για τους φοντιστές. Αυτές οι ευέλικτες διευθετήσεις μπορεί να σημαίνουν εξ αποστάσεως κατοίκων εργασία, ευέλικτα ωράρια σε δόσεις μέσα στη μέρα ή μείωση του συνόλου των ωρών εργασίας. Το δικαίωμα αυτό για τις ευέλικτες διευθετήσεις είναι δικαίωμα να ετηθεί κανείς τέτοιες ευέλικτες διευθετήσεις για σκοπούς φροντίδας εφόσον θέλει να είναι φροντιστής κάποιος. Οι εργοδότες οφείλουν να λάβουν υπόψη και να αποκριθούν σε αυτές τις αιτήσει, ε, αιτιολογώντας οποιαδήποτε άρνηση. Αυτό μπορεί να είναι ένα προσωρινό δικαίωμα, η διάρκεια του μπορεί να είναι ε, αντικείμενο εύλογου περιορισμού που θα ε, αποφασίζουν τα κάτι μέλη και αν η διάρκεια περιοριστεί, τότε υπάρχει δικαίωμα επιστροφής την αρχική διευθέτηση για την εργασία στο τέλος της συμπεφωνημένης περίοδου. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα, λόγου χάρη εάν υπάρχει αλλαγή στις συνθήκες. Μείωση του χρόνου εργασίας δεν χρειάζεται πια, οπότε ο εργοδότης πρέπει να λάβει υπόψη το αίτημα, την αίτηση, ή η επιστροφή στη θέση εργασία σε ανάλογη θέση και με βελτιώσεις ενδεχομένως. Εάν δεν υπάρχει περιορισμό στη διάρκεια. Υπάρχει μάλιστα απαγόρευση για τη διοικητική μεταχείριση εφόσον απλώς και μόνο γίνει έτοιμα, αίτηση για να λάβει κανείς άδεια και άρνηση για τα ευέλικτες διευθετήσεις. Επίσης υπάρχει προστασία από απόλυση ή ε, μη ευνοϊκή μεταχείριση, εφόσον κάποιος ζητήσει απλώς ευέλικτες διευθετήσεις στην εργασία του. Το βάρος της απόδειξης σε περίπτωση απόλυσης είναι παρόμοιο με τα ζητήματα ισότητας βάσης του κοινωτικού δικαίου. Λίγο πολύ αυτή είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόμενη. Θα ήθελα σύντομα να αποτιμήσω την πρόταση αυτή. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου. Να την καλωσορίσουμε. Λόγω του ρόλου των ανδρών, κατά κύριο λόγο, ο οποίος ενισχύεται, Ελαμβάνει άλλη ε, προβολή ως προς την ε, γονική, την άδεια πατρότητας. Επίσης η άδεια των φροντιστών είναι πολύ σημαντική. Δεν υπάρχει σωρά τα κατημέλη και για τις σοβαρές ασθένειες ή τους εξαρτώμενους συγγενείς, τα εξαρτώμενα μέλη. Η αμοιβή κατά τη διάρκεια της άδεια είναι σημαντική. Τα δικαιώματα αυτά επίσης είναι εξατομικευμένα και η ευελιξία που μπορεί να καλύψει ανάγκες ε, των εργαζομένων με ευθύνε φροντιστών είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, επόμενη, η οδηγία για την εγκυμοσύνη και την πατρότητα παραμένει απαράλλαχτη. Εάν δούμε λοιπόν τις ελλείψεις, υπάρχουν κάποιες εξεπλάγει που δεν υπάρχει καμία αμνία στο προήμιο της σύμβασης για την εξάλληψη των διακρίσεων κατά των γυναικών του ΟΗΕ. Μια πολύ σημαντική σύμβαση από αυτήν την έννοια, ιδίω το πρέμιό τη. Ακόμη και αν δεν έχει ε, κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω τα περισσότερα κάτι μέλη ε, πρέπει να την ε, εφαρμόσουν, ιδίω αυτή τη διάταξη. Και όλος ιδιαίτερο το ψήφισμά σα του Σεπτεμβρίου 2016 αναφέρει αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέω, αναφέρει και τονίζει το ρόλο των στερεοτύπων των δύο φύλων σε ζητήματα εξισορρόπησης οικογενειακού επαγγελματικού βίου. Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση και απέτηση να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα αυτά στο άρθρο 5 της σχετικής σύμβασης. Οι άδειε είναι αρκετά σύντομες, ιδίω αυτή των φροντιστών. Αν έχει κάνει μια σοβαρή ασθένεια στην οικογένειά σου, δεν φτάνουν πέντε μέρες. Προσωπική εκτίμηση αυτή, αλλά για το δικαίωμα να ετηθεί κανεί ευέλικτε εργασιακέ διαθετήσει. Είναι κάπω αδύναμο. Έχει δικαίωμα κανεί να ετηθεί, αλλά δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει. Δεν είναι ισχυρό αυτό το δικαίωμα. Ούτε μπορεί να κάνει κάτι μακροπρόθεσμα, μπορεί μόνο προσωρινά να μειώσει τι ώρε εργασία του. Πολύ σημαντικό επίση, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τη νομική βάση, δεν υπάρχουν καθόλου συνέπειες για τα δικαιώματα που εγείρονται στην ε, κοινωνική ασφάλεια, είτε βάση καταστατικού ε, ή τα, ε, τα δικαιώματα βάσει της εργασίας. Αυτό εμένα μου φαίνεται κάπως. Ας δούμε τι ε, θα σημαίνει η πρόταση αυτή αν εγκριθεί, όπως τώρα είναι διαμορφωμένη, για τις κατοχώρες. Η άδεια πατρότητα ε, στι κατοχώρε είναι δύο μέρε πληρωμένε. Μπορεί κανεί να πάρει μέρο τη γονική άδεια ε, για τρει μέρε, αλλά χωρί να πάρει χρήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα βήμα πρόοδου με τη συγκεκριμένη πρόταση τη Επιτροπή. Δεν έχουμε καθόλου πληρωμένη γονική άδεια εκτό από τι συλλογικέ συμβάσει στη δημόσια δίκηση. Κάποιε συλλογικέ συμβάσει επίση σε άλλου τομεί, αλλά γενικώ δεν πληρώνονται. Εδώ λοιπόν θα έχουμε πληρωμένη άδεια που είναι και αυτό ε, πρόοδος. την άδεια των φροντιστών, στις κάτω έχουμε περισσότερες δυνατότητες. Δέκα μέρες το χρόνο πληρωμένη άδεια κατά 70% του ελάχιστου μισθού, οπότε δεν αλλάζει τίποτα και έχουμε και μακροπρόθεσμη άδεια φροντιστού, μία αμοιβόμενη έξι εβδομάδες. πολύ χαμηλότερο γιατί υπολογίζονται ώρε ανά εβδομάδα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για τι κατοχώρε είναι ότι η ομάδα για την οποία μπορεί κανεί να παρέχει φροντίδα δεν είναι απλώ συγγενή και οικογένεια, είναι πολύ ευρύτερο ορισμό. Είναι όλε οι κοινωνικέ σχέσει. Μπορεί να είναι κάποιο ο οποίο πραγματικά έχει άμεση ανάγκη βοήθεια και να είναι απλό γείτονα. Δεν αναγκαίνει να είναι και συγγενή εξαίματο. Ως προς την ευέλικτη εργασία στις κάτω χώρες έχουμε πολύ πιο προηγμένη νομοθεσία, διότι έχει δικαίωμα να προσαρμόσει κανείς τις ώρες εργασίας του για κάποιες περιόδους, αλλά και τον συνολικό αριθμό ώρων που δουλεύει. Έχει επίσης το δικαίωμα να προσαρμόσει το πρόγραμμά του και Ιδίω αν δουλεύει σε εταιρεία με περισσότερου από 10 εργαζομένου. Ω προ το σύνολο των ορών εργασία, ο εργοδότη πρέπει να δεχτεί το αίτημα προσαρμογή των ορών εργασία και του χρόνου εργασία, εκτό εάν υπάρχουν σοβαροί επιχειρησιακοί λόγοι που να το εμποδίζουν. Πρέπει δηλαδή να γίνει δεκτό το αίτημα. Οι λόγοι άρνηση μπορεί να είναι σοβαρά διοργανωτικά προβλήματα. Ως προς το ε, ωράριο εργασία την εβδομάδα υπάρχουν περισσότερε δυνατότητε άρνηση, γιατί πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση των συμφερόντων του εργαζομένου και του εργοδότη. Ω προ τον εργασιακό χώρο, το δικαίωμα αίτηση είναι ίδιο και παρόμοιο τέλο πάντων με αυτή την πρόταση τη Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Κάποια συμπεράσματα. Η οδηγία είναι κάπως αποσπασματική Δηλαδή ανακαλείται άδεια για την, η οδηγία για την, οδηγία, για την γονική άδεια, εάν περάσει αυτή. Υπάρχει σχετική συνοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ε, προσέγγιση της με άλλες οδηγίες και, άλλες, και άλλα νομοθετήματα, αλλά μέχρι ενός σημείου υπάρχει αυτή η συνοχή. Διότι δεν συμπεριλαμβάνεται η άδεια μετρότητας. Εκεί μας λείπει λίγη συνέπεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το ότι υπάρχουν πληρωμένε άδειε πλέον, άδειε για του φροντιστέ και ευέλικτε εργασιακέ διαθετήσεις και όλο ιδιαίτερο εντό του πλαισίου που έχει σκιαγραφηθεί ε, από την αρχή τη παρουσιασή μου. Η φροντίδα είναι ένα πολύ σοβαρό ε, ζήτημα, ιδίω σε μια κοινωνία με την ε, υπερχείρανση του πληθυσμού. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πάμε και παραπέρα με τις 10 δράσεις εάν λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες για τη φροντίδα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η τελευταία διαφάνεια. Thank you very much, ε, Ευχαριστούμε πολύ την ε, καθηγήτρια Μπάρη για την παρουσίαση. Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον ε, δόκτωρα Τίμο Αντίλα από το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Γεβασκυλά στη Φιλανδία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω το λόγο σε αυτό το σημαντικό εργαστήριο και να σας μιλήσω για την έρευνά μας. Η δική μου ομιλία αφορά, αφορά λοιπόν περισσότερα την ε, εμπειρική μα έρευνα και ο σκοπός είναι να εξετάσουμε πώς ο εργάσιμο χρόνος συνδέεται με την ε, εξισορρόπηση του εργάσιμου και του γυναικού χρόνου και επίση θέλουμε να δείξουμε ε, την ποικιλομορφία που υπάρχει μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά τον εργάσιμο χρόνο. Και θα παρουσιάσω το, τα τελευταία δεδομένα σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό προσκήνιο. Αρχικά, ο εργάσιμο χρόνο ε, ε, αποτελεί όλο και περισσότερο ένα σημείο εστίαση για την ανάλυση και τη συζήτηση ό,τι αφορά την απασχόληση. Ε, υπάρχει μεγάλη αλλαγή προς ε, την μεταβιομηχανική οικονομία ως μοντέλο με βάση τη γνώση, με πιο ευέλικτο εργάσιμο χρόνο και ο εργάσιμος χρόνος είναι βασική μεταβλητή. Από την μεταβιομηχανική ε, κατηγορία, το μεταβιομηχανικό μοντέλο εργάσιμου χρόνου, αυτό σημαίνει ότι έχουμε την ρύθμιση των ε, συλλογικών ε, προτύπων και διαφοροποίηση του χρόνου και των προτύπων ε, και αυτό σημαίνει ότι κάπως ε, δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς μεταξύ του εργάσιμου και μη χρόνου πια. Επόμενο διαφάνεια. Ο εργάσιμο χρόνο ε, και η ευελιξία δύσκολα συνδυάζονται με αυτή την ισορροπημένη ζωή. Η ευελιξία συνήθω ε, δεν αποβαίνει πέρα ε, του οικογενειακού χρόνου ή του προσωπικού χρόνου ζωή και πάντα θα πρέπει να πιέζουμε για περισσότερη τέτοια ισορροπία. Συνήθως ε, η ευελιξία αυτή αξιοποιείται από τους ε, εργοδότες ε, για να επιβάλλουν έτσι, κακά ωράρια στους εργαζομένους τους και ούτε καθεξής. Όταν εξετάζουμε τον χρόνο εργασίας, συνήθως επικεντρωνόμαστε σε μία ξεχωριστή πτυχή διάσταση του εργάσιμου χρόνου. Συνήθως ε, μιλούμε για τον αριθμό των ωρών, τον χρόνο δηλαδή. Όμως όταν έχουμε μία ευρύτερη προσέγγιση, καταρχάς έχουμε την χρονική και τη χωρική ευελιξία, Αυτές οι δύο διαστάσεις, κατά τη γνώμη μας, διαμορφώνουν ε, ε, ένα πρότυπο και έτσι οδηγούμαστε και στις διαφορές μεταξύ των επιμέρους χωρών. αλλά και οι ομάδες των εργαζομένων διακρίνονται με βάση αυτό το κριτήριο. Σε ό,τι αφορά την χρονική ευελιξία, εννοούμε την διάρκεια, το χρονισμό, δηλαδή κακές, δηλαδή ε, κακά ωράρια, αρνητικά ωράρια, ρυθμός, διαρρυθμός εργασίας, όλο ένα και πιο σημαντική αυτή η πτυχή στην ε, πράξη αυτού σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας και ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η αυτονομία είναι σημαντική από τη διάσταση από αλλά και επειδή ε, κάπως αντισταθμίζει τις αρνητικές ε, συνέπειες ε, των διαβριμένων ωραρίων, των αντικοινωνικών ωραρίων όπως αναφέρονται και της πίεσης χρόνου. Χωρική ευελιξία σημαίνει εργασία εξ αποστάσεως, ταξίδια και Κάποια αποτελέσματα τώρα από τις τελευταίες μελέτες για τις ε, εργα... συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε ε, τις συνεντεύξεις από 37.000 εργαζομένους στην Ευρώπη. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στον χρόνο εργασίας και στην ε, ε, συμφιλίωση του εργάσιμου και προσωπικού βίου. Το ερώτημα είναι ε, πώς, ε, πόσο καλά θεωρείς ότι συνδέονται και συνδυάζονται η ε, προσωπική σου ζωή με τις υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις. Και υπάρχει μια διαβάθμιση από το 1 μέχρι το 5. Εδώ έχετε λοιπόν έναν ευρωπαϊκό χάρτη, βλέπετε την αναλογία των απαντήσεων που έχουν πολύ θετικέ απαντήσεις και εύκολα βλέπετε τα αποτελέσματα. Δεν φαίνονται τόσο καθαρά τα χρώματα, αλλά ουσιαστικά με τα πιο σκούρα χρώματα βλέπετε τα πιο θετικά αποτελέσματα, με την καλύτερη δηλαδή ισορροπία και εδώ στο χάρτη βλέπετε την διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Στις σκανδιναβικές χώρες, ιδίως ε, ε, στη Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, είναι πολύ θετικές απαντήσεις. Περίπου η μισή ε, απάντησαν ότι η εργασιακή του ζωή συνδυάζεται πολύ καλά με την προσωπική του ζωή. Μετά έχουμε κάποιες χώρες της κεντρικής Ευρώπης που επίσης έχουν θετικά αποτελέσματα, Αυστρία, Τσεχία και το καθεξής. και κάποιες πιο φιλελεύθερες ε, χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία ε, και εδώ έχουν ε, θετικές απαντήσεις. Από την άλλη πλευρά έχουμε κάποιες χώρες της Νότιας Ευρώπης, Πορτογαλία, Ιταλία, όπου κάτω από το 1 τέταρτο των απαντήσεων είναι θετικές. Το σημερινό εργαστήριο αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση. Και αν δείτε τα ποσοστά απασχολησιμότητας ε, των γυναικών στην Ευρώπη, ε, τα ανώτερα τέτοια ποσοστά ε, τα βρίσκουμε στη Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Κατοχώρες, Φερλανδία, Ηνωμένα Βασίλεια και Αυστρία. Αν δείτε στον χάρτη, Υπάρχει ε, σημαντική συσχέτιση μεταξύ του, της ε, συμφιλίωσης προσωπικής και εργασιακής ζωής ε, και της απασχόλησης των γυναικών. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τα συμπεράσματα εδώ έχουμε πέντε βασικά μοντέλα, το υπηρετικό, το βρετανικό, το ανατολικό, το νότιο και το σκανδιναβικό. Βλέπουμε ότι το σκανδιναβικό και το φιλελεύθερο έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής. Μετά θα δούμε τη διαφοροποίηση που υπάρχει στον εργάσιμο χρόνο μεταξύ των μοντέλων αυτών βάσει της δικής μας ε, ενοιολογικής προσέγγισης διακρίνουμε διάφορες πτυχές ε, του εργάσιμου χρόνου, την διάρκεια, τον χρονισμό, τον ρυθμό, την αυτονομία και την ευελιξία στον χώρο εργασίας. Εδώ βλέπετε λοιπόν πώς ε, διαφοροποιούνται αυτές ε, οι πτυχές του εργάσιμου χρόνου. Για παράδειγμα, στο σκανδιναβικό μοντέλο, αν πάρουμε αυτό το μοντέλο σαν ε, σημείο αναφοράς, βλέπετε ότι έχουμε αντικοινωνικές ώρες ή κακά ωράρια τέλος πάντων κάτω από το μέσο όρο. Ε, καλή αυτονομία, καλός ε, ρυθμός και βαθμός πίεσης και υψηλός βαθμός ευελιξίας ό,τι αφορά το χώρο εργασίας. Αυτό το μοντέλο λοιπόν μας δίνει την ε, καλύτερη ισορροπία μεταξύ ε, εργασιακής και προσωπικής ζωής μπορούμε να το συγκρίνουμε με το ανατολικό μοντέλο που έχουμε μεγαλύτερα ωράρια, λιγότερη αυτονομία. ή μπορούμε να συγκρίνουμε το σκανδιναβικό με το νότιο μοντέλο, όπου αυτά τα κακά ωράρια αρνητικά είναι ε, πιο συχνά και υπάρχει και πάλι χαμηλός βαθμός αυτονομίας. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, όπου συνοψίζονται τα συμπεράσματά μας και βλέπετε πώς ε, συνδυάζονται όλε αυτέ οι πτυχέ του εργάσιμου χρόνου με την αίσθηση που έχει κανεί για την ισορροπία μεταξύ προσωπική και εργασιακή ζωή. Εδώ βλέπετε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κόκκινη μπάρα, τόσο ε, πιο αρνητικά είναι τα αποτελέσματα. Επομένω, ε, Αυτά τα κακά ωράρια εργασία έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο. Ε, η μεγαλύτερη αυτονομία έχει θετικό αντίκτυπο. Η πίεση χρόνου μειώνει την αίσθηση της ισορροπίας μεταξύ εργάσιμου και προσωπικού βίου. Και εδώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σημασία ε, της ευελιξίας σε ό,τι φορά το χώρο εργασία και πώς συνδυάζεται με αυτή την αίσθηση. Και αυτό είναι κατανοητό. Όσο μεγαλύτερη ευελιξία υπάρχει προς το χώρο εργασία. τόσο και πάλι αυτό επηρεάζει την αίσθηση ισορροπίας. Από προηγούμενες μελέτες προκύπτει ότι υπάρχει διαφορά εδώ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες αξιοποιούν την ε, κατοίκον εργασία για να συγκεντρωθούν πραγματικά στη δουλειά τους, ενώ οι γυναίκες ε, για να ασχοληθούν ε, με ζητήματα που έχουν να κάνουν την οικογένεια. Συμπερασματικά, είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο ο εργάσιμος χρόνος. Πρέπει πάντα να θέτουμε το ερώτημα για ποιον, ε, ποιον εξυπηρετεί αυτή η ευελιξία και έχουμε βρει σημαντικέ διαφορέ μεταξύ αυτή τη ισορροπία εργάσεων και προσωπικού βίου ανάλογα με τη χώρα και τα μοντέλα. Ε, ξέρουμε ότι και η νομοθεσία και οι συλλογικέ διαπραγματεύσει ε, επηρεάζουν ε, αυτό το φαινόμενο, καθώ και οι ε, διαφορές διαφορέ τη αφορά τον ε, χρόνων εργασία και τι σχετικέ συμπεριφορέ. Κοινωνικοί κανόνε συνήθω ορίζουν ε, ποιος ε, δικαιούται αυτή την ευελιξία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much, ε, doctor. Σας ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρα Τίμο Άντλη, για την πανδική σας παρουσίαση και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην δόκτωρα Κωνσταντίνα Δαβάκη. good afternoon, everyone. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Δυστυχώς, επειδή είμαι η τελευταία ομιλήτρια, και έχουμε δύο πάρα πολύ διακεκριμένων ομιλητών που κάλυψαν πολύ έδαφος. Θα αναγκαστώ να αλληλεπικαλύψω κάποια από αυτά που είπαν πλέον. Δεν το είχα προβλέψει. Η σχέση δημογραφικών πολιτικών με τις πολιτικές ε, συμφιλίωσης κοινωνικού, επαγγελματικού βίου ήταν και το θέμα μιας ε, μελέτης που διενέργησα για την Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Θα καλύψω και κάποιες άλλες διαστάσεις ε, πάντως. Περάστε με διαφάνεια αν μπορείτε. Άλλη μία. Μάλλον λείπει η εισαγωγή μου από ό,τι φαίνεται. Α, εδώ είμαστε. Ευχαριστώ. Το δημογραφικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, τεκμηριώνεται με βιβλιογραφία. Τρεις κρίσεις βιώνουμε παράλληλα, την οικονομική, τη δημογραφική κρίση και την κρίση των προσφύγων. Στη μελέτη μου καλύπτω και το μεταναστευτικό, αλλά δεν ε, είναι της παρούσης. Η γονιμότητα πλήττεται από τις τομικές συνθήκες αλλά και από τις οικογενειακές, οικογενειακές και πολιτικές απασχόλησης. Επηρεάζεται επίσης από συμπεριφορές, από τις πολλές και διάφορες αναπαραγωγές τεχνολογίες και τα θεσμικά και τις θεσμικές ρυθμίσεις. Πέφτουν τα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν υπάρχει σχέση αιτίου ατού ξεκάθαρη, τουλάχιστον μεταξύ του βαθμού της κρίσης και της τάσης γονιμότητας. Για παράδειγμα, μεταξύ των μέτρων λιτότητας που πλήττουν τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, στην Ελλάδα, βλέπουμε αναστροφή της ε, κατάστασης γονιμότητας, αλλά στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, δεν βλέπουμε κάποια συσχέτιση προς τον παρόν και καταλαβαίνετε έτσι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι οι μεμονωμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαρόκη συμπεριφορά. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί η καθολική εκκλησία να επηρεάζει για την περίπτωση Πορτογαλίας αλλά και της Ιταλίας Και γι' αυτό δεν ε, μειώθηκαν τα ποσοστά γονιμότητας πολύ. Έχουν γίνει και εμπειρικές μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ απασχόλησης, α, μάλλον ανεργίας και ποσοστών γονιμότητας. Δηλαδή οι άνεργοι ε, επηρεάζονται τι αποφάσει τη περιγονιμότητας από την έλλειψη εργασίας, που είναι και λογικό. Από την άλλη πλευρά, κάποια κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικογενειακέ πολιτικές. Πιο πολιτικές περισσότερης συμπερίληψης που βοηθούν και δείχνουν και τι αλλαγέ στι οικογενικέ δομέ. Για την Ουγγαρία, παραδείγματο χάρη, η οικογένεια ξεκολουθεί να ορίζεται ω ζευγάρι τεροφιλόφιλο με παιδιά. Βέβαια, είναι σημαντικό να δούμε και κατά πόσον ε, τη γονιμότητα επηρεάζουν και οι μη παραδοσιακέ οικογενειακέ πολιτικέ, όπω η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία και η συμμετοχή των ανδρών περισσότερο στη φροντίδα. Βλέπουμε ότι συνήθω στις χώρες που προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη γονιμότητα με περιγενικές πολιτικές, τελικά η διάκριση είναι πιο ισοβαρής μεταξύ των δύο μελών, μεταξύ δύο γονέων. One before, yes. Thank you. Um, recent research in... Πρόσφατη έρευνα σε 24 χώρες δείχνει ότι όσο το πλαίσιο είναι πιο προοδευτικό προς την ισότητα, τόσο πιο ίση είναι και η διάκριση σε ό,τι αφορά τη μη αμοιβόμενη εργασία. Επίσης αυξάνεται των 900 στην αγορά εργασία. Όχι και πολύ βέβαια, αλλά αυξάνεται. Τα υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας πάντοτε είναι αποτέλεσμα μεγαλύτερης ισορροπίας ε, μάλλον πολιτικών που πράγουν την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματική ζωής. Επίσης η αλλαγή ρόλων και η πιο σοβαρή κατανομή των ε, καθηκόντων φροντίδας σχετίζεται με τις ε, καλύτερες συνθήκες για την ισορροπία γυναικής πραγματικής ζωής. Εδώ αναφέρω και την πράσινη βίβλο για την αντιμετώπιση δημογραφικών αλλαγών που έχει ήδη καλυφθεί από κάποια προλαλήσαντα. Είναι μια σύσταση αυτή τη πράσινη βίβλου άξιση αύξηση τη γενική απασχόληση. Από το 2007 και μετά είχαμε πολιτικέ λιτότητε σε πολλέ χώρε τη Ένωση. Και τα μέτρα αυτά είχαν αρνητικέ επιπτώσει, ιδίω στον Ευρωπαϊκό Νότο. Υπάρχει επισφάλεια στη γενική απασχόληση. Και αυτό αυξάνει την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια. Και είναι κατανοητό ότι κάποιες συνθήκες μπορεί να μην έχουν επηρεάσει ακόμα κάποιες χώρες ό,τι αφορά τα ποσοστά γονιμότητας, αλλά σύντομα θα το κάνουν. Το δε σημαντικότερο είναι πως επηρεάζεται πολύ σοβαρά η συμβιλίωση οικογενειακής επαγγελματικής ζωής. Ανεξαρτήτως του αν μιλάμε για παραδοσιακή οικογένεια, για μονογονικές οικογένειες ή άλλες διευθετήσεις οικογενειακές. Γιατί όμως σχετίζονται οι πολιτικές ε, της συνοικής απασχόλησης και πόσο βοηθούν ε, την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και εγκληματικής ζωής. Υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα στις διάφορες χώρες ε, και μεγάλο, μεγάλη βιβλιογραφία, διαφορετικές ταξινομήσεις και τυπολογίες Και αυτό στο οποίο θα επιμείνω είναι αυτό που θεωρώ ότι είναι η ισορροπία εργασιακού και οικογενειακού βίου. Δηλαδή πώς ε, υπάρχει μια ισορροπημένη κατανομή προτεραιοτήτων μεταξύ των ατομικών δραστηριοτήτων και της ζωής που περιλαμβάνει ψυχή, προσωπική ανάπτυξη κτλ. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη πως η αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών του φίλου και του νοικοκυριού, τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, η οικογενειακή και εργασική πολιτική και το κατά πόσο υπάρχει συμφιλίωση ή δεν υπάρχει συμφιλίωση με την ε, μία αμοιβόμενη εργασία, αυτά προσδιορίζουν και καθορίζουν την ισορροπία μεταξύ οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Το 2015 Φερνάντες ε, Κρεχόιτ, ή κάπω έτσι προφέρεται, δεν ξέρω ακριβώ. και συνάδελφοι διενέργησαν μια μελέτη και έχουν καταρτήσει έναν δίκτυ για το work-life balance. Βλέπουμε ότι στη Δανία και Σουηδία είναι στην κορυφή, Σλοβακία και Ελλάδα ουραγή. Υπήρξαν κάποιες ε, κριτικές παρατηρήσεις ό,τι αφορά την ισορροπία οικογενειακής πνευματικής ζωής, μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά δεν αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα. Κυρίως τη μεσαία τάξη. Αν θέλουμε όμως να έχουμε πολιτικές συμπερίληψεις, Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλή απασχόληση. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα εργα... Ε, δεδομένα, στοιχεία. Αν θέλουμε να χαράξουμε πολιτικές που θα εξασφαλίζουν για όλους ισορροπημένη οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Δεν θέλω να με για τις άδειες, γιατί ακούσαμε μια καταπληκτική παρουσίαση προηγουμένως για τα θέματα αυτά. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη πως όταν μιλάμε για άδειε, είναι ένα κεντρικό εργαλείο πολιτικής, αλλά πάντοτε πρέπει να μας απασχολεί το επίπεδο της αμοιβή, πόσο καλό είναι. Πρέπει να δούμε επίσης τη διάρκεια και το δικαιούχο. Γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις. Για εγγύους δεν θα μιλήσω γιατί τις καλύπτει οδηγία για την γονική άδεια. Για να δω όμως τι θέλω να πω εδώ. Άδεια φροντιστών. Θέλω να προσθέσω κάτι γιατί ακούγοντας ε, την παρουσίαση σκέφτηκα πως αυτό το βήμα είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αλλά διερωτώ με αν το δημογραφικό στοιχείο αν μπορούμε να δούμε τη διαφορά μεταξύ άδεια φροντιστών και γονική άδεια. Και τη σαφή συσχέτιση με τις δημογραφικές προτεραιότητες. Και αν δούμε τι γίνεται για τη γονική άδεια με την οδηγία τη σχετική και πώς έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, ένα πάρα πολύ καλό βήμα προς και όλοι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την εξέλιξη. Αλλά αν τα συγκρίνουμε με το τι γίνεται για του φροντιστέ, βλέπουμε ότι δεν έχουν γίνει πολλά γιατί δεν υπάρχει συσχέτιση με το μέλλον τη Ευρώπη, με τη νέα γενιά. Μιλάμε για το βάρο, για το ηλικιωμένου που αντιμετωπίζονται έτσι. Και ε, νομίζω ότι αυτό είναι ντροπή. Και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για του φροντιστέ. Για έναν απλό λόγο, ότι οι Ευρωπαϊκή Πολιτεία δεν είναι γονεί. Υπάρχουν και πολλοί ανήπαντροι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φροντίζουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μπορεί να μην είναι παιδιά κατά ανάγκη. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα της συσχέτισης δημογραφικών και γενικών πολιτικών ή της μη συσχέτισης. Επόμενη διαφάνεια. Υπηρεσίες παιδικής φροντίδας. Αυτονόητο είναι ότι υπάρχει ανάγκη. Με την άδεια μπορεί πρώτον δεν είναι επαρκή η άδεια, δεύτερον μπορεί να μειώσει τη συμμετοχή των γυναικών, να είναι επιζήμιε δηλαδή άδειε, ε, αν είναι ιδίω μακροχρόνιε και δεν. Βλέπουμε και κάποια μέτρα για τον επιμερισμό των βαρών. Ε, οι υπηρεσίες λοιπόν πρέπει να υπάρχουν. και έχει αποδειχθεί από ένα σκανδιναβικό, με το σκανδιναβικό παράδειγμα, το ότι αυτές οι διευθετήσεις και η ύπαρξη των λόγω υπηρεσιών, η παροχή των λόγω υπηρεσιών έχουν βοηθήσει τα μάλα συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε επίσης και τα αποτελέσματα του αντίθετου, δηλαδή της μείωσης, της περικοπής ε, υπηρεσιών, πόσο αυτό βλάπτει τη συμμετοχή των γυναικών. Επόμενη διαφάνεια. Η εργασιακή ευελιξία είναι δίκοπο μαχαίρι. Δίνει αυτονομία και έλεγχο από τη μία, αλλά έχει και κάποια αντίθετα αποτελέσματα. Επηρεάζει ε, τη σχέση μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής. Οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερη ευελιξία, είναι πιο παραγωγικοί, δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ να ανακυκλωθούν σε κάποια άλλη θέση. Η τεχνολογία επίσης βοηθάει. Απ' την άλλη πλευρά όμως ε, κάνει πιο ασαφή τα όρια μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής. δεν ορίζεται ξεκάθαρα το που αρχίζει και που σταματάει η δουλειά. Και κάποιο πρέπει να είναι πάρα πολύ αποφασισμένος και πεθαρχημένος για να έχει μια ισορροπία. Επίσης η κουλτούρα της θέσης εργασίας επηρεάζει ε, τη χρήση των ευέλικτων μορφών εργασίας. Μπορεί να είναι άτακτες οι ώρες εργασίας και αυτό μπορεί να διαταράξει και τις δραστηριότητες των γυναικών στην αγορά εργασίας λόγω αυτής της φροντίδας, της έμφυλης φροντίδας. Η ευελιξία μπορεί να είναι επιζήμια όταν η μητέρα πρέπει να πάει να πάρει το παιδί από το σχολείο. προωθούνται τελικά οι ετεροφιλόφιλες παραδοσιακές ε, οικογένειες και οι ανάγκες ε, για την ε, ισορροπία εργασίας και οικογενειακής ζωής, αλλά υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές επιθυμίες. Οι νέοι μπορεί να αργήσουν να σχηματίσουν οικογένεια. Ή κάποιοι πιο ηλικιωμένοι μπορεί να θέλουν να παραμείνουν πιο πολύ στην αγορά εργασίας και με την ευελιξία μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Και η ιδεολογία, ο πολιτισμός, η κουλτούρα επηρεάζουν τη στάση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, δεν τους έχει δοθεί απαιτούμενη προσοχή. οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά έχουν επηρεάσει επίσης ε, τις διαφορετικές ε, κοινωνικές ε, πολιτικές και όχι μόνο ατομικές προτιμήσεις. Υπάρχει λοιπόν ανομοιογένεια της μη εργασία. εργασίας με βάση τη φιλετική εθνική καταγωγή, την τάξη κτλ. Τέλος, κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Η λογική πίσω από την ισορροπία οικογενειακής επαγγελματικής ζωής είναι ε, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Να υπάρχει βιωσιμότητα και του κράτους πρόνοιας. Η γονιμότητα σχετίζεται και με οικονομικούς παράγοντες και την ε, ασφάλεια της ε, απασχόλησης, αλλά και με την, τον εκμερισμό εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας. Υπάρχει σημαντική ε, διακύμανση των εθνικών πολιτικών για το work-life balance και οι στάσεις και οι ρόλοι δεν έχουν προσεχθεί τόσο πολύ. Θα πρέπει να δίνουν περισσότερη βάση στην ε, ισότητα των δύο φύλων σε ό,τι αφορά την ισορροπία οικογενειακής και ζωής και να ενθαρρύνουν ένα νέο μοντέλο για τους ε, πατέρες και ελπίζω με την μονάδια πατρότητα αυτό να βελτιωθεί. Επίσης θα πρέπει στις πολιτικές να αναγνωρίζετε και να λαμβάνετε υπόψη η ε, ποικιλομορφία των αναγκών και των συνθήκων. Και οι πιο ε, επιτυχημένες πολιτικές είναι αυτές που θεωρούν το άτομο και ως άτομο που κερδίζει κάποιο εισόδημα, αλλά και ως ένα άτομο που φροντίζει κάποιο άλλο μέλος οικογένεια και αυτό κυρίως στις σκανδιναβικές ε, χώρες πολιτεία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις μορφές ανισότητα. Όχι τις ηλικέ μόνο. Τις περιορισμένες ευκαιρίες, περιορισμένες δυνατότητε και πώς αλληλεπικαλύπτονται. Επίση θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των γυναικών. Τέλος. Και ο ίδιος όρο αυτό αυτος αυτός, work-life balance, βάζει την εργασία πρώτα. Work. Είναι ώρα όμως και ελπίζω να έρθει αυτή η ώρα σύντομα να δοθεί έμφαση στη δεύτερη συνιστόσα, life, στη ζωή δηλαδή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρα Δαβάκη, για την παρουσίασή σας. Και τώρα να δώσω τον λόγο στα μέλη για τη συζήτηση, κυρία Μλίνερ. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο. Πρώτα απ' όλα πάρα πολύ ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για αυτή την τόσο διεξοδική επισκόπηση. Θα χρειαστεί χρόνος για να αφομοιώσω τις λεπτομέρειες. Πολύ ενδιαφέρον ε, αυτό το σεμινάριο και οι συνάδελφοι στις εθνικές μας βουλές θα είχαν κάθε λόγο να κάτσουν να ακούσουν αυτά που υπόθηκαν. Απλώς μερικές αντιδράσεις. Για σας κυρία Δαβάκη. Περισσότερο από όλα όσα είπατε, στα οποία θα προσυπέγραφα ευχαρίστω, μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε στο τέλο. Η δουλειά, κατά τη δική μου άποψη, δεν έπρεπε να είναι αντίφαση ω προ τη ζωή, να αποτελεί αντίφαση. Δεν Έπρεπε να είναι μέρο τη ζωή. Είναι λε και προσπαθούμε να ορίσουμε τα πράγματα αρνητικά. Λε και πρέπει κανεί να προασπιστεί τη, τη ζωή του. Είμαι πεπισμένη ω άνθρωπο ότι θα είμαι πιο χαρούμενη εάν έχω επιλογή. Την δυνατότητα να αξιοποιήσω όλα μου τα ταλέντα. Το να κερδίζει κανείς λεφτά δεν είναι κακό. Μου άρεσε πολύ λοιπόν η προσέγγιση σας όταν είπατε ότι οι γυναίκες που είναι μέρος της αγοράς εργασίας έχουν πιο ικανοποιητική ζωή. Και αυτό λένε και οι ίδιες. Συμφωνώ λοιπόν πλήρως με την ιδέα που συμπεριλαμβάνεται στο Σύνταγμα των Πολιτειών να επιδιώκουμε την ευτυχία. Εδώ χρειάζεται μια κοινωνική αλλαγή και νομίζω ότι το είπατε όλοι πολύ ξεκάθαρα σήμερα. Τέλος πάντων στις ομιλίες σας. Μπορεί να δημιουργήσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής αυτό θα ήταν μια ωραία επιδίωξη. Ευχαριστώ κύριε Μπλίνερ. Θέλετε να απαντήσετε τώρα. Ναι, αν μπορώ. Πολύ ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Να ξεκαθαρίσω ότι η δουλειά μπορεί να είναι τρομερά ικανοποιητική. Ως γυναίκα που εργάστηκα όλη μου τη ζωή, από τότε που απεφύτησα, ξέρω τι είναι να έχει κανείς μια δουλειά από τον Δεν ξέρω αν θα έλεγα το ίδιο αν ήμουν σε μια σύμβαση μηδενικών ωρών. Ακριβώς το σχόλιο σας αυτό έρχεται να επιρρώσει αυτό που είπα. Όταν μιλάμε για εξισορρόπηση επαγγελματικού οικογενειακού βίου, μιλάμε για την μέση τάξη, έτσι, ως έννοια Αυτή ήταν και η επίκριση που δεχτήκαμε στην βιβλιογραφία για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και βίου. Δεν είναι μια επιδίωξη που όλοι θα υποστηρίζαμε. Στην πολιτική όταν ορίζουμε την έννοια, αλλάζουν τα πράγματα. Αν θέλουμε λοιπόν να συμφιλειώσουμε την επαγγελματική ζωή και τον ιδιωτικό βίο, αυτό είναι ένα στοιχείο. Αλλά οι πολιτικές σε επίπεδο ε, χάραξης πολιτικής είναι κάτι το διαφορετικό. Οπότε ναι, είμαι βεβαία, εάν είχα μια σύμβαση με δενικών ορών, δεν θα ήμουν και τόσο πάρα πολύ χαρούμενη και θα ανησυχούσα για το μέλλον μου, για να μην σας πω και για την επιβίωσή μου. Δεν θα είχα καμία ισορροπία, πιστεύω. Αλλά συμφωνώ, όταν κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες του, τα ταλέντα του, μπορεί με την παιδεία, την εκπαίδευσή του, να φτάσει να ευχαριστιέται τη ζωή του, αυτό ακριβώ είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των πολιτικών μα. Η δική μου ευχή είναι αύριο οι γυναίκες με συμβάσει μηδενικών ωρών να μπορούν σε 12 μήνε να πούν αυτό που είπατε κι εσεί: ότι μπορούν να είναι χαρούμενες και να μιλήσουν για την πολιτική εξισορρόπηση επαγγελματικού οικογενειακού βίου. Uh, uh, Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Μαχτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις, τους τεκλημένους μας για τις τρεις ομιλίες τους. Ε, συνολικά, όσα μας είπατε, και το λέω και στους τρεις, ε, θέλω να πω το εξής. Είμαι άνδρας και αν αλλάξει η δουλειά μου και πρέπει να, δουλάξω, να δουλέψω βράδυ, δεν με νοιάζει καθόλου. Εάν πρέπει να δουλέψω νωρί το πρωί, σκασίλα μου. Ε, το ίδιο και για τα Σαββατοκύριακα. Αν ήμουν ε, γυναίκα, θα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Είμαι άντρα, είμαι εδώ στι Βρυξέλλε, τέσσερι μέρε τη βδομάδα. Αν ήταν η γυναίκα μου στη θέση μου, δεν θα ήταν τόσο εύκολο. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη και τι πολιτικέ μα, για να είμαστε αξιόπιστοι, για να είμαστε ε, πιστική σε αυτό που προτείνουμε, ε, πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Ε, να σα δώσω ένα παράδειγμα τον εαυτό μου. Είμαι μεγάλο, αλλά είμαι πατέρα πρόσφατα. την περασμένη εβδομάδα, την περασμένο χρόνο μάλλον, ζήτησα άδεια πατρότητα ακριβώ λόγω του μωρού και μου είπαν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό στη χώρα μα. Είμαστε λοιπόν συνομοθέτε, αλλά εδώ είμαστε σαν το χωριό το γαλατικό του Αστερίξ. Δηλαδή κάνουμε αυτά που θέλουμε για τους άλλους και δεν ισχύουν για μας. Και το εξή να πω ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη κατά κάτι μέλη πρέπει να λάβουν μια οριστική απόφαση, μια τελεσίδικη απόφαση για τη θέση που θέλουμε να δώσουμε στις γυναίκες στην κοινωνία μας. Να σταματήσουν οι υποκριτικές ε, στάσεις. Ε, δείτε τι είπατε προηγουμένως. Είπα τα διαμετρότητας, πατρότητας κλπ. κλπ. ότι έχουμε μια προσέγγιση βάση του φύλου, αλλά έχουμε στην πολιτική μα χάραξη βάση του φύλου. Γιατί έχουμε Επιτροπή Γυναικών εδώ, υπάρχει Επιτροπή Ανδρών, γιατί υπάρχει Επιτροπή Γυναικών. Γιατί ακόμη συνεχίζουμε να αγνοούμε τι θέση ακριβώ θέλουμε να δώσουμε στι γυναίκε στην κοινωνία μα. Όταν μιλάμε για τη γυναίκα στο δημόσιο χώρο, οι γυναίκε είναι θύματα των ε, ε, παρενοχλήσεων. Δείτε τι γίνεται με την παρουσία τη γυναίκα στον χώρο τη εργασία. Το είπατε και εμένα και ΔΕ. Διαφορά στου μισθού. Δυσκολίε εξισορρόπηση προσωπική και επαγγελματική ζωή. Το είπατε, όταν μια γυναίκα θέλει να ε, δουλέψει στο σπίτι είναι επειδή θέλει να ε, φροντίσει την οικογένεια. Όταν ένα άντρα θέλει να δουλέψει στο σπίτι είναι για να συγκεντρωθεί καλύτερα. Όταν μιλάμε για του μισθού, όταν μιλάμε για την πολιτική γεννήσεων. Ε, ε είναι πάντοτε οι γυναίκε στο κέντρο τη συζήτηση. Εδώ κάνατε τρεις παρουσιάσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά νομίζω το πρόβλημα των πολιτικών μας θα πρέπει να επικεντρωθούν στα δικαιώματα των γυναικών, ισότητα ανδρών και γυναικών και ούτω καθεξής. Ε, είπαμε, θέση της γυναίκας ε, από εδώ και από εκεί πρέπει να το δούμε ως κάτι συνολικό. Διότι θα καθόμαστε αιώνες να μιλάμε για τη θέση της γυναίκας, αν δεν λάβουμε μια απόφαση. Θα είμαστε εδώ στην Επιτροπή Γυναικών. Εγώ θα χαρώ πολύ μια μέρα να μην υπάρχει πλέον αυτή η Επιτροπή Γυναικών. Δεν θα έχουμε πλέον αυτή την προσέγγιση βάση του, ήλου, του φίλου. Δεν είναι το ίδιο μια γυναίκα και ένα άντρα Αυτό δεν μα απασχολεί, αλλά δεν πιστεύετε ότι Βεβαίω χρειάζεται νόμοι, χρειάζεται εδώ το κίνητρο των νόμων, τη νομοθεσία, αλλά δεν ε, χρειάζεται, πιστεύετε, επειδή κάνατε τη διαφορά μεταξύ σκανδιναβικών χωρών και του Νότου, για λόγου που αναφέρατε προηγουμένω και πολύ σωστά του απαριθμίσατε. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι η νομοθεσία πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση και τον ε, πολιτισμό, του παιδεία. Για να πάψει να τίθεται το ερώτημα από την πρώτη στιγμή που γίνεται κανεί, Ποιο είναι ο ρόλος της μικρής μου αδερφή, ε, της φίλης μου, της γυναίκας μου, της μαμάς μου και το καθεξής. Δεν ξέρω αν ήμουν σαφή στην παρουσίασή μου. Νομίζω ότι οι καλύτεροι νόμοι να εγκριθούν, παρόλα αυτά θα υπάρχει ε, μια ομάδα ανδρών με, ε, των 50 ετών με κουστούμι και χραβάτα που θα παίρνουν αποφάσεις για τις γυναίκες. Και όχι το ανάποδο. Και δεν είμαστε στο τέλος αυτής της ιστορίας. Διάβαζα πρόσφατα δημοσιεύματα που εξηγούσαν ότι είναι σημαντική η νόμη, αλλά εάν δεν υπάρξει ε, εκπαιδευτική πολιτική, πολιτική πολιτιστική, θα παραμείνουμε ουραγοί και ουραγοί των ουραγών. Από τις τρεις παρουσιάσεις που κάνατε, παρά τις καλές προθέσεις που εξαγγέλλονται από εδώ και από εκεί, εάν αύριο περάσει εδώ ένα νομοσχέδιο, σε αυτό το κοινοβούλιο, σε αυτό το κοινοβούλιο το ευρωπαϊκό, διότι και εδώ έχει πολύ υποκρισία και φαρεσιασμό, Πιστεύω ότι θα εξλαγούμε δυσάρεστα από το αποτέλεσμα τη ψηφοφορίας. Δεν είμαι καν βέβαιο ότι όσα τα είπατε, μόλι μα είπατε εδώ, θα τα δεχτούν κάποιοι από του Ευρωπαίου εδώ. Ότι ναι, συμφωνούμε και από αύριο πρέπει να υπάρξει ισότητα. Απόλυτη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οπότε α πάψει υποκρισία, α τα δούμε όλα μαζί από κοινού και να βεβαιωθούμε ότι αυτή η Επιτροπή χρειάζεται να εξαλειφθεί, να μην χρειάζεται. Και ότι η ισότητα ισχύει ε, διατομεακά σε όλους τους χώρους, σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαχτά. Να δώσουμε τώρα το λόγο και πάλι στους εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν. Well, thank you very much. Not, not more than minutes. Ε, για τρία λεπτά έκαστος παρακαλώ. Τρία λεπτά για να λύσουμε αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστά μιλήσατε για τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εμείς εξετάζουμε μόνο μία πτυχή εδώ. Και εντός αυτής της ε, μίας πτυχής, της ισορροπίας δηλαδή προσωπικού και εργάσιμου βίου, εξετάσαμε την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Ένα από τα στοιχεία που ε, αναφέρθηκαν σήμερα είναι ότι πρέπει να δώσουμε και κίνητρα στου άντρε. Αυτό είναι κάτι το καινούριο. Αλλά βέβαια δεν φτάνει. Η κουλτούρα μας ε, ακολουθεί τα ανδρικά πρότυπα εντό αγωγικών. Βέβαια, αυτό το βλέπουμε παντού. Και τα σημεία που δείξατε σίγουρα έχουν να κάνουν και με αυτό. Το σχόλιο της κυρίας Δαβάκη επίσης είναι πολύ σημαντικό από αυτή την άποψη. Έχουμε ένα συγκεκριμένο φίλτρο και τρόπο σκέψης και είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε ε, τι ακριβώς προσφέρουν οι επιμέρους πολιτικές ε, στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Και γι' αυτό μίλησε για τις ε, άδειες μεταποδοχών. Βέβαια αυτό δεν είναι το παν, ούτε η ευελιξία στον εργάσιμο χρόνο είναι το παν. Πρέπει να αλλάξουν πολλά ακόμα. Υπάρχει σεξισμός σε πολλούς τομείς του ανθρώπινου και ιδιωτικού βίου. Όμως υπάρχουν ορισμένες ε, πρωτοβουλίες, για παράδειγμα η γαλλική πρωτοβουλία ε, μια συγκεκριμένη καμπάνια ε, σεξίσμου σε genre. Αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένε δομικέ αντιλήψει ω προ τον ρόλο του άντρα για τη Γυναίκα και δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα αυτά σε τρία λεπτά. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε δομές, τρόπους σκέψης, μοντέλα συμπεριφορών και ε, ανισομέρεια στις ε, σχέσεις εξουσίας. Ναι, και εκπαίδευση βεβαίως. Αλλά δεν φτάνει. Σαφώς και η παιδεία συνιστά σημαντικό βήμα αλλά δεν φτάνει. Uh, yes, uh... Μάλιστα. Αντίλα. Συμφωνώ σε πολλά από τα όσα είπατε. Μιλήσατε για διαφορές ε, μεταξύ χωρών. Αναφερθήκατε στις ε, σκανδιναβικές χώρες διαφορές μεταξύ ορισμένων χωρών συνδέονται στενά και με, το, με την οικονομική δομή και τις δομικές αλλαγές ε, της οικονομίας. Το εργατικό δυναμικό, για παράδειγμα, στη Σκανδιναβία έχει υψηλή μόρφωση και ξέρουμε ότι οι ευέλικτες πρακτικές επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες ομάδες εργαζομένων. Για παράδειγμα, για τους υψηλά ιστάμενους αυτό σημαίνει μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας. για να προσδιορίσει ο κάθε εργαζόμενος πότε εργάζεται και πότε όχι. Ε, για όσους έχουν χαμηλότερες θέσεις, για παράδειγμα αυτό μπορεί να σημαίνει ε, αρνητικά ωράρια ή διαβριμένο ωράριο και τα καθεξής. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τις διαφορές μεταξύ διαφορών ε, ομάδων εργαζομένων και τις ε, συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται, γιατί εκεί εντοπίζονται τεράστιες διαφορές. Και νομίζω ότι αυτές οι διαφορές είναι ακόμα πιο σημαντικές ε, από τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κύριε Ταβάκη, Ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί σας. Όπου σταθώ και που βρεθώ, αυτό λέω, ότι πρέπει να υπάρχει ολιστική προσέγγιση. Μόνο λοιπόν αν εξετάσουμε ένα πρόβλημα ολιστικά, μόνο εάν εξετάσουμε τις διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους πολιτικών και δεν τις εξετάζουμε μεμονωμένα. Μόνο τότε λοιπόν μπορούμε να έχουμε και αποτελέσματα. Σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο, στην ισορροπία μεταξύ εργάσιμου και προσωπικού βίου, γιατί αυτό ήταν και το θέμα σήμερα, υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει ο νομοθέτης και στην παρέμβαση τον ιδιωτικό βίο που ορίζει, για παράδειγμα, τις αναπαραγωγικές επιλογές και το Αυτό μπορεί να κάνει ο νομοθέτης. Και εδώ πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές χώρες. δεν υπάρχουν οι ίδιες αξίες ή τα ίδια κοινωνικά μοντέλα απαραίτητα. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε την ε, ε, πολυμέρεια αυτή. Γι' αυτό ο νομοθέτης θα πρέπει ε, να θεσπίσει τις υπηρεσίες αυτές που θα δώσουν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες στους πολίτες για να αξιοποιήσουν τη μόρφωσή τους, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να δώσουν λοιπόν τη δυνατότητα στους πολίτες μέσω των υπηρεσιών αυτών να ε, πάρουν αυτόνομα και τελείως ελεύθερα αυτές τις αποφάσεις που θα τους ε, ευχαριστήσουν. Μέχρι να γίνει αυτό όμως και παρότι είμαι φιλόδοξη, δεν θεωρώ ότι ε, θα επιτευχθεί σύντομα η ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Μέχρι τότε λοιπόν χρειαζόμαστε την επιτροπή αυτή, την κοινοβουλευτική επιτροπή. Ωστόσο, θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχή εάν ε, τα πράγματα βελτιωνόνταν τόσο, τόσο πολύ που τελικά ε, θα ήταν παροχημένη αυτή η επιτροπή. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Και τώρα κυρία Μόνικα καλημέρα. Πολύ σύντομα ένα σχόλιο Νομίζω ότι και η ιστορία είναι όπως την έχουμε ζήσει όλες αυτές τις γενιές ε, χαραγμένη από τους άνδρες και καλό θα ήταν να μην έχουμε μόνο αντρική ιστορία, his story αλλά και her story. Uh, Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και το Ιδρυματικό Τμήμα ΓΑΜΑ για την διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου. Uh, Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία, παρακαλώ, γιατί τη συνάλληψη λίγο. Πέντε λεπτά. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, είστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει τις κάρτες ψηφοφορία. Το σημείο 5 λοιπόν της Μέσης Διάταξης είναι εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατικής για την Αναπηρία. Έγκριση του σχεδίου θέση μορφή τροπολογιών. Η εισηγήτριά μας είναι η κυρία Ρόζα Σταράς Φεραγκούτ. Ξεκινούμε λοιπόν την ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογίες από 24 έως 28 μπορούμε να τις ψηφίσουμε από κοινού. Συμφωνείτε? Ωραία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. εγκρίνονται. Τροπολογία 79. Έχουμε μια προφορική τροπολογία εδώ. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρόπο 29. Α, όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 31. Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Το 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Καλά δεν τα λέω. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε από κοινό από τη 36 έως τη 38. Όχι. Καλώς. 36. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπλή 42 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι περ. Κατά αποχές, να ελέγξουμε παρακαλώ έρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολέγη 44, ψήφι περ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45, ψήφι περ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47, ψήφι περ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολία 52. Ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουν παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 63 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Από την 68 έως την 74 να ψήσουμε, όχι. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίφθηκε. Την 71 θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Μάλιστα. Ε, 73 τώρα. Ψήφι υπέρ. Υπέρ. 73. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. 76 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Κάθε φορά το ίδιο αποτέλεσμα. 77 υπέρ, κατά, Αποχές. Συνάδελφοι, πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 78. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, ρωτώ, μπορούμε να ψηφίσουμε από την 1 έως την 5 από κοινού. Ωραία, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 8, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εντάξει, να ελέγξουμε αν θέλετε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 με προφορική τροπολογία. Ε, υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψήφι υπέρ. Α, η Μάλιν κάτι θέλει να πει. Ναι, συγγνώμη. Θα τα πω αγγλικά. Γιατί τις ε, έστειλε πολύ αργά κύριε Κωνσταντής Κακούνεβα τις τροπολογίες. Μιλάει για άτομα με αναπηρία και ιδίως ε, γυναικών και κοριτσιών. Για να είμαστε πιο συνεπείς Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία. Στη 12. Πρέπει να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία καταρχάς. Την δεχόμαστε την προφορική υπέρ, κατά, αποχές,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 με προφορική τροπολογία, ναι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε την 20, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 21 ψήφι κατά, ποχές, εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ και την εισηγήτρια. Επόμενη συνεδρίαση, 25 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι. Μην το ξεχάσετε. Και τώρα στις 5 Ξεκινάει η συνεδρία των συντονιστών. Καλό απόγευμα στους υπολείπους.